τροπολογίες περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Ε, πρέπει επίσης να σας ενημερώσω ότι οι δηλώσεις ε, επί της ε, ψήφου για αυτήν την ψηφοφορία θα υπάρξουν στην επόμενη Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Δηλαδή δεν θα έχουμε τώρα χρόνο για επεξηγήσεις ψήφου. Και περνάμε τώρα ε, σε αυτά που στις τροπολογίες τεσσάρων πολιτικών ομάδων Έχουμε καταρχήν την ε, ε, τροπολογία υπαριθμών 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Περνάμε τώρα, μισό λεπτό, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα απορρίφθηκε λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 14 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 27, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εδώ πράγματι χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτό. Δεκτή η τροπολογία. Πάμε τώρα στην υπαριθμόν 15, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Παράγραφος 2, τροπολογία υπαριθμών 4, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία και περνάμε στην 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 18 υπέρ κατά αποχές. Εδώ πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική επαλήτευση, η οποία και άρχεται. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Απορρίπτεται η τροπολογία. Και περνάμε τώρα στο αρχικό, στο πρωτότυπο κείμενο, σε τρία τμήματα, ψηφίζουμε σε τρία τμήματα, τα δύο πρώτα τμήματα είναι χωρί ονομαστική ψηφορία υπέρ του πρώτου παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεκτό τρίτο ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία δεκτό δεκτή τροπολογία. Πάμε στην παράγραφο 3, ε, τροπολογία υπαριθμών 19, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην παράγραφο υπαριθμών 4, τροπολογία 5, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 5, τροπολογία 6, υπέρ παρακαλώ, κατά απορρίπτεται. Η 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο μάλλον πάμε μετά την παράγραφο 5, η τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7, τροπολογία 21, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα στην παράγραφο 9, τροπολογία υπερθμών 8, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης απορρίπτεται. Η 31, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το αρχικό κείμενο ποιος είναι υπέρ του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 9 η τροπολογία υπαριθμών 23 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω ότι είναι σαφές το αποτέλεσμα αλλά τέλος πάντων ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην παράγραφο, μετά την 10, η 24 παρακαλώ, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ του αρχικού κειμένου, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η 32 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται αρχικό κείμενο της ε, παραγράφου 12 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ηλεκτρονική επαντήθευση για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε ψηφοφορία απορρίπτεται και περνάμε τώρα στην τροπολογία υπεριθμών 16 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται η παράγραφος 13, ε, μετά την 13 η 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και η 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία υπερτιμών 10. Εδώ υπάρχει μία προφορική τροπολογία του κυρίου Μέσσερ Σμιτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εκ μέρου του ECR θέλω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία που αλλάζει την τροπολογία με την έννοια ότι διαγράφεται το δεύτερο τμήμα, άρα αυτό που λέει based on inaptitude, language, hostility κτλ. Αυτά δηλαδή που αφορούν την εχθρότητα έναντι του Ηνωμένου αυτό διαγράφεται. Και το μόνο που απομένει και από αυτού ψηφίζουμε είναι προ την παρέτηση του ε, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Γιούγκερ. Αυτό παραμένει. Πρόεδρος, έχετε αντιρρήσει από αυτού. Αν έχετε αντιρρήσει πρέπει να σηκωθείτε. 40. 40 βουλευτές ε, έπρεπε να σηκωθούν για να δείξουν την ε, αντίθεσή τους. Σηκώθηκαν πολύ περισσότεροι, άρα απορρίπτεται η τροπολογία σας. Ψηφίζουμε για την αρχική μορφή της τροπολογίας υπέρ, κατά, αποχές, Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Απορρίφθηκε οριακά. Πάμε τώρα στις τροπολογίες 1 και 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται η τροπολογία 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεκτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Και περνάμε τώρα στο ψήφισμα, στο σύνολό του, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Εγκρίνετε το ψήφισμα. Τα πρακτικά αυτή της συνεδρίασης, κύριε και κύριοι, θα υποβληθούν στην επόμενη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου προς έγκριση. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα ε, θα υποβάλω στα ε, όργανα, στους θεσμούς που αναφέρονται στο ψήφισμα. Διακόπτεται λοιπόν η, ε, η περίπτωση Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λύεται η σημερινή συνεδρίαση.